Allora, iniziamo i lavori della Commissione. Να ξεκινήσουμε τι εργασίε τη Επιτροπή. Ε, συνεχίζουμε τι εργασίε που διακόψαμε σήμερα το πρωί και συνεχίζουμε από το σημείο 22. Αναφορά 1845 του 2013 του Ρολάντ Έγκερ, Αυστριακού υπηκόου, με 14.658 υπογραφές για την ευρωπαϊκή ασφάλιση, για την αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων σε πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία σύμφωνα με τον αναφέροντα δεν συμμορφούνται ε, με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ο αναφέρον είναι παρόν, θα του δώσουμε το λόγο για πέντε λεπτά για να μας ε, παρουσιάσει το θέμα της αναφοράς ομολογώ ότι ε, είμαι λίγο μπερδεμένος. Λέγομαι Ρόλαντ Έκε, όχι αυτός που είπατε. Ε, εκπρόσωπος του Ράιλαντ Τούρεκ είναι εκεί μπροστά, ο κύριος που φοράει τώρα τα ακουστικά. Okay, so, um, Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ διότι μας δώσατε την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Φίλοι της γης στην Ευρώπη ιδρύθηκε ο φορέας μας ε, λίγο μετά τα τραγικά μετά της ε, Φουκουσίμα τον Μάρτιο του 2011. Τότε ε, απαιτήσαμε εδώ και τώρα να κλείσουν οι εγκαταστάσεις όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων υψηλού κινδύνου στην Ευρώπη. Και είπαμε να μην δοθεί παράταση ζωή και στις παλαιές εγκαταστάσεις, ούτε να κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις. Επίσης, απαιτήσαμε κάποιο είδου ε, νομική δέσμευση για το κλείσιμο όλων των ε, εργοστασίων παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2020 και επίσης απαιτήσαμε να σταματήσουν τα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων προς την πυρηνική βιομηχανία και είπαμε να σταματήσει η Ευρώπη να στηρίζει ε, και την χρήση πυρηνική ενέργεια. Επίση, ζητήσαμε βιώσιμε και αηφόρε επενδύσει για ανανεώσιμε μορφέ ενέργεια και για ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τι έγινε έκτοτε. Ο πυρηνικό κλάδο στην Ευρώπη κατάφερε να φέρει τούμπα τα πράγματα για όλε τι εγκαταστάσεις να πείσουν ότι είναι ασφαλεί. Αυτό είναι εξόχω. Ε, μάλλον είναι οίκιστα πιστικό μετά την Φουκουσίμα, γιατί ξέρουμε ότι η φιλοσοφία του 100% ασφάλεια είναι τελείως ε, λάθος, γιατί δεν, δεν, στέκει. Και είναι σαν να μην έγινε ποτέ η καταστροφή στην Φουκουσίμα, οπότε πάρα και αυτοί οι 800.000 του οποίους εγώ εκπροσωπώ, σαν να μην υπάρχουν ποτέ, θεωρούμε ότι σε πάρα πολλές χώρες έχουμε επικίνδυνε εγκαταστάσει οι οποίε μπορεί να πάρουν παρά τη ζωή και το οποίο για μα είναι απαράδεκτο. Οι βασικέ μα προσπάθειε τώρα επικεντρώνονται στο να ενημερώσουμε τον κόσμο, να το ειδικοποιήσουμε και να έχουμε ε, ενεργειακέ μορφέ ενέργεια, να πείσουμε την κυβέρνηση και να σταματήσουν οι κυβερνήσει να επιδοτούν και να κατασκευάζουν νέε πυρηνικέ εγκαταστάσει όπω θέλουν όπως ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχουμε πολλά θέματα τα οποία κρεμούν ε, όσον αφορά την ποινική ενέργεια, έχουμε και όλα αυτά τα σοβαρά ατυχήματα. Και θέματα σχετικά με τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται εκεί. Έχουμε μια μελέτη που δημοσιοποιήθηκε ε, στην Βιέννη από ένα τεχνικό ε, Ινστιτούτο ε, πριν από δύο εβδομάδες λοιπόν και λέει ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και θα, πρέπει να έχουμε ανάπτυξη των ανανεώσιμων. Οπότε σας παρακαλώ υποστηρίξτε τον απαλλαγή Ευρώπη από τον πυρηνικό κίνδυνο η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε και τώρα. Ο λόγος την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Άταλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον αναφέροντα για την εισήγησή του. Σας παραπέμπω στο άρθρο 194 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζει αυτό το άρθρο ότι στην ενέργεια τα νέα μέτρα δεν επιδρούν το ενεργειακό μείγμα της κάθε χώρας. Επομένως δεν έχουμε αρμοδιότητα να αναλάβουμε δράση όσον αφορά τα κράτη-μέλη και τις ποινικές τους εγκαταστάσεις. Πέραν τούτου, πάντως η ποινική ασφάλεια για την Επιτροπή είναι θέμα προτεραιότητα και γι' αυτό και κατόπιν του ατυχήματος του Φουκουσίμα αντιδράσαμε άμεσα. Πήραμε εντολή από, την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάναμε τεστ αντοχής παντού στην Ευρώπη, ε, Τρει φάσεις έγινε αυτό. Πρώτα-πρώτα κάποιο είδου αυτοαξιολόγηση από αυτού που έτρεχαν τα εργοστάσια. Επίση, είχαμε από τι εθνικέ κάποιες αρχέ κάποιε εκθέσει ε, αξιολόγηση από ισοτήμου και μετά ελέγξαμε τα κράτη-μέλη σε σχέση με το, ε, με, με το τι είχε αξιολογηθεί ότι πρέπει να βελτιωθεί. Ε, όλα αυτά επομένως πέρσι τα ξαναεξιολογήσαμε και κάναμε μια έκθεση όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης μας έδωσε εντελή να αναθεωρήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά και επί τη βάση των συμπερασμάτων που αντλήσαμε από το ατύχημα της Φουκουσίμα και των τεστ αντοχής δημοσιοποιήσαμε αυτήν την, ε, την πρότασή μας για μια οδηγία ε, πυρηνικής ασφάλειας ανεξάρτητους, ε, ε, ανεξάρτητες δημιουργικές αρχές, ε, προτείνουμε διαφάνεια, να έχουμε ενωσιακού, πανενωσιακούς στόχους, να είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας, να αντιδράσουμε και να έχουμε αξιολόγηση ισοτήμων παντού, επί τη βάση των αρίστων πρακτικών και μηχανισμούς, ούτως ώστε να υπάρξουν κάποιες καθηγητές γραμμές για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι ε, εναρμονισμένες Τώρα όσον αφορά τις νέες εγκαταστάσεις πρέπει να επενθυμίσουμε ότι αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό γίνεται υπό την εποπτεία των εθνικών δημιουργικών αρχών. Παρόλα αυτά η πρότασή μας εισάγει το ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια ε, επιθεώρηση αυτών των εγκαταστάσεων και επίσης ζητούμε ε, να υπάρχουν επιθεωρήσεις ασφαλείας όποτε κλείνει ο κύκλος ζωής μιας ποινικής εγκατάστασης και υπάρχει θέμα παράτασης της ζωής αυτής της εγκατάστασης. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Έγινε ένα μικρό λάθος ανταλλάξαμε τις αναφορές, διότι ξεκινήσαμε με την αναφορά υπαρχημών 22. Mm. Εγώ είχα δώσει το λόγο στον ε, κύριο Έγκερ. Και για την αναφορά 23 ακούσαμε τον κύριο Ούλριχ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευτυχώς ε, κατάφερε να συνοψίσει και τα δύο θέματα τα οποία τέθησαν. Η αναφορά υπαριθμών 22 θέτει το θέμα της ενιαίας ασφάλισης για τα πυρηνικά ατυχήματα, ε, ενώ το θέμα της αναφοράς παριθμών 23 του κυρίου Ούλριχ είναι η αναφορά που καλεί για αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ε, κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας, επικρίνοντας και το παρόν σύστημα. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σατάρτ, μας παρουσίασε συνολικά και τα δύο θέματα για την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το τι κάνει. Έκανα διευκρίνηση για τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο, διότι αυτή τη στιγμή θα συζητήσουμε από κοινού και τα δύο θέματα. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Άουκεν. Just... Κυρία Πρόεδρε, ζητώ πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όλο αυτό το θέμα της ασφαλίσεως για αυτό το λόγο σταμάτησε η πυρηνική ενέργεια στη Δανία. Βέβαια, προηγήθηκε πρώτα μακρά συζήτηση με πολύ αξιόπιστες πληροφορίες Όμως είχαμε προχωρήσει πολύ με όλη την ομοθεσία να έχει εγκριθεί και μετά άρχισε η συζήτηση γιατί θα γινόταν εάν ας πούμε συνέβαινε ένα μεγάλο πυρηνικό ατύχημα σε ένα μεγάλο πυρηνικό σταθμό στην Σουηδία, κοντά στα σύνορα με τη Δανία. Και μετά διαπιστώσαν ότι η πυρηνική βιομηχανία ποτέ δεν θα μπορούσε να αντασφαλιστεί. Καμιά μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία δεν δεχόταν να την αντασφαλίσει. Αυτές οι επιχειρήσεις, ξέρετε, το μυρίζονται το χρήμα. Αν λοιπόν ήταν πράγματι η πυρηνική ασφάλεια τόσο ασφαλής, όσο, η πυρηνική συγγνώμη, ενέργεια, τόσο ασφαλής όσο λένε, ό, θα έχει όλες τις ασφαλείς που χρειάζεται. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα έπεισε και το κοινό στη Δανία αλλά και την δανική κυβέρνηση ότι καλύτερα να δούμε τι λένε αυτοί που ξέρουν από λεφτά. Και εφόσον αυτοί που ξέρουν από λεφτά δηλαδή δεν τολμούν να ασφαλίσουν τους πυρηνικούς σταθμούς, τότε μάλλον φαίνεται ότι ίσως καλύτερα να μην αναλάβουμε και εμείς οι ίδιοι τον κίνδυνο. Έτσι επιχειρηματολόγησαν δηλαδή. Και έτσι δεν προχώρησε η νομοθεσία για τα πυρηνικά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι ευθύνη και τη Κομισιόν. Όπως είπατε και εσεί ο ίδιο ε, σας απασχολεί η πυρηνική ασφάλεια και δίνεται μεγάλη προτεραιότητα και άλλα μπλα μπλα που μας είπατε. Ίσως λοιπόν ενδιαφέρον για σας και θα μπορέσετε να με πείσετε τουλάχιστον εμένα, αν μου εξηγήσετε για ποιο λόγο εσείς γνωρίζετε περισσότερα περί ασφαλείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αν υποτίθεται ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος και έτσι και αυτοί δεν πρόκειται να χάσουν τα λεφτά τους. Ε, ποιες είναι οι σκέψεις σας όμως για την ασφάλεια. Και γιατί δεν ασφαλίζουν τα πυρηνικά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ιραδα, Ιραδα Μπαμπαλτιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά έχουμε συζήτηση για τα πυρηνικά ζητήματα εδώ στην Επιτροπή μας. Από τότε που έχω έρθει όλο το ίδιο συζητάμε και ανέκαθεν έλεγα ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ενέργεια του παρελθόντος και όχι ενέργεια του μέλλοντος όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Πρόκειται για μια ενέργεια η οποία δημιουργεί περιτούς κινδύνους για το μέλλον, διότι υπάρχουν προβαλή, προβλήματα όπως το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς επίσης και τα προφανή ατυχήματα σε πυρηνικά εργοστάσια και οι συνέπειές τους. Υπάρχει το πασίγνωστο ε, παράδειγμα της Ευρώπης ε, στο Τσερνομπίλ και αυτή τη στιγμή τόσο ε, το να ζητούμε ασφάλιση ε, για τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πυρηνικά εργοστάσια. Είναι σίγουρα μια ε, καλή άγουσα για να περικόψουμε λίγο τις, τα όσα κάνει αυτή η βιομηχανία που όπως έλεγα είναι η ενέργεια του παρελθόντος και φυσικά είναι και ένα αποτελεσματικό αντισύστημα σε κάποιο βαθμό. Επιπλέον, Υπάρχει ένα εργοστάσιο, το Σάντα Μαρία, το οποίο ζητούν να κλείσει αμέσω. Ένα εργοστάσιο το οποίο είχε ξεκινήσει με τι ευχέ όλων, υπήρχε ενδιαφέρον από την ε, κυβέρνηση της Ισπανίας ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένανε να ξεκινήσει τη λειτουργία του στο εγγύς μέλλον. υπάρχουν πάρα πολλά παροχημένα εργοστάσια, όπως για παράδειγμα αυτό του Σάντα Μαρία και υπάρχει και το αίτημα για πυρηνικοποίηση, ε, για ε, διαφορετικό ενεργειακό μείγμα και ζητάτε να υπάρχει πυρηνική ενέργεια σύνδεξης αλλά υπάρχει και το αίτημα η πυρηνική ενέργεια, ε, κυρίως η πυρηνική ενέργεια σχάσης, να ε, γίνει ενέργεια του παρελθόντος το συντομότερο δυνατό. Ελπίζω να τηρηθούν οι υποσχέσεις του εγγύης ε, μέλλον. Ελπίζω και η υπόσχεση για την πυρηνική ενέργεια σύνδεξης να μπορέσει να υλοποιηθεί σύντομα. Θεωρώ όμως ότι ε, αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον της ανθρωπότητας και θέλουμε να δώσουμε ένα καλό μέλλον για τα παιδιά μας, θα πρέπει να κλείσουμε τους πυρηνικούς σταθμούς το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλισης, είναι ε, κατά την άποψή μου μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε ζητώ ήδη από την αρχή την κατανόησή σας, διότι για την πορεία της συνεδριάσεως θα παρακαλέσω, έστω και αν απάντησε η Κομισιόν για δύο αναφορές, δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει λόγο να μην μπορέσει να παρουσιάσει ο ένας αναφερόμενος την δική του αναφορά. Γι' αυτό παρακαλώ να, να δοθεί ο λόγος στον αναφερόμενο της αναφοράς 1845 που ε, λόγω της συγχύσεως τελικά δεν μπόρεσε να παρουσιάσει την αναφορά του. Παρακαλώ να του δοθεί η ευκαιρία. Το θέμα αυτό της ημερησίας διατάξεως δεν έχει εκφωνηθεί. Ζητώ συγγνώμη που τα θέτω αυτά και πάλι. Μιλώ για την 1845. Έδωσα το λόγο στον αναφερόμενο. Και ο ίδιος μου είπε ότι προτιμά να μιλήσει αυτός. Μα ήταν ο σωστός άνθρωπος. Είστε ο κύριος Ρόναντ Μπέγκερ. Σας έδωσα το λόγο και είπατε όχι, να μιλήσει αυτός. Με συγχωρείτε να σα διακόψω. Δώσατε το λόγο στον Ράινχαρτ Ούλρικ και κοιτάξατε εμένα. Και αναφέρατε... Όχι. Ίσως να μην με ακούσατε καλά. Διότι εγώ έδωσα το λόγο σε εσά. Ανέφερα την αναφορά σας, μίλησα για την αναφορά σας, έδωσα το λόγο σε εσά και εσείς παρετηθήκατε. Αλλά βεβαίως έχετε το λόγο, έχετε το δικαίωμα να λάβετε το λόγο. Νόμιζα ότι ήταν δική σα επιλογή να μην μιλήσετε. Δεν είναι πρόβλημα για μένα. Μπορείτε να πάρετε το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να πω λίγα λόγια για την σημαντική αυτή αναφορά για την ευθύνη από πυρηνικά ατυχήματα. Αγαπητοί κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μετά από την ήδη αναφερθήσα ατυχή περίπτωση της Φουκουσίμα είναι καθαρό ότι τα, οι ζημιές από πυρηνικά ατυχήματα ανέχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ε, δολαρίων ή ευρώ το μέγα μέρος της ζημίας βαρύνει τελικά το κοινό. Το σύστημα που ακολουθούν είναι ότι είναι περιορισμένη η ευθύνη τους εξ αρχής. Οι διεθνείς συμφωνίες που συνήφθησαν μετά Παρισίων, Βιέννης και ούτω καθεξής προβλέπουν περιορισμένη ευθύνη για την βιομηχανία, για, την, για τον φορέα της βιομηχανίας. Η πυρηνική ε, βιομηχανία έτσι έλαβε ένα σημαντικό προνόμιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζημιών που με κανένα τρόπο δεν είναι πλέον δικαιολογημένο. Ο Επίτροπος Έτιγκερ κατ' επανάληψη ζήτησε αυξημένη ευθύνη για τους ε, πυρηνικούς σταθμούς και είπε καθαρά ότι πολλές Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι αυτό που θέλουν δηλαδή πολλοί Ευρωπαίοι είναι, όπως είπε ο για το 2012 τον Οκτώβριο, είπε εντολή μου δεν μπορεί να είναι να κάνω φτηνό το ρεύμα από πυρηνική ενέργεια με dumping αποζημιώσεων. Στο, κάθε, στο, στο τέλος της γραφής και ο κάθε οδηγός αυτοκινήτου οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη για ατυχήματα προκαλεί. Φαίνεται πάντως τώρα ότι έχει ανακρούσει πρίμνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν προτείνει πλέον παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το 2012 γαλλική μελέτη καταλήγει ότι σε ενδεχόμενο μεγάλο πυρηνικό ατύχημα στην Ευρώπη μπορεί να φτάσει η συνολική ζημιά μέχρι 400 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 400 φορές παραπάνω από το ποσό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο απογοητευτικό είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει οδηγία για τη ρύθμιση της ευθύνης από πυρηνικό ατύχημα, ούτε κανονισμό, σχεδιάζει μοναχά μια απλή ανακοίνωση. Ανακοίνωση για μας είναι ένα ιδιαίτερα αδύναμο μέσο που θέλει τώρα να προτιμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν δίνει κανένα ξεκάθαρο μήνυμα απαντώντας στις καταστροφικές συνέπειες της Φουκουσίμα. Ευχαριστώ. Κύριε Τάτ, θέλετε εσείς να ε, προσθέσετε κάτι. Να διευκρινίσω ότι στην προηγούμενη παρέμβασή μου δεν αναφέρθηκα στο θέμα της ασφαλίσεως. Αναφέρθηκα μονάχα στα θέματα που θέτει στην αναφορά το προηγούμενο αναφερόμενο. Για τούτην εδώ την αναφορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να επαναλάβει ότι δέχεται την συμμετοχή όλων των stakeholders σε αυτή τη συνεχιζόμενη συζήτηση για υποχρεωτική ασφάλιση των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη και ιδίως βέβαια τα θέματα που θέτει η κοινωνία των πολιτών. Η αναφορά είναι όντω επίκαιρη, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκύψει το θέμα ήδη από το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, έχει κάνει ε, μελέτη με νομική γνωμοδότηση για την ευθύνη για αποζημίωση τρίτων, καθώς και έχει ομάδες εμπειρογνωμόνων που έχουν, ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συναντηθεί έξι φορές μέχρι τώρα. Και τον Ιούλιο 2013 μέχρι τον Οκτώβριο έκανε και σχετική δημόσια διαβούλευση. Η έκβαση της διαβούλευσης δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη συνένεση για να ρυθμιστεί το θέμα της ευθύνης των πυρηνικών σταθμών απέναντι σε τρίτους. Οι περισσότεροι που συμμετέσχαν στις δημόσιες διαβουλεύσεις συμφωνούν με τους αναφερομένους ότι πρέπει να υπάρξει κάλυψη της ευθύνη έναντι τρίτων και η μεγάλη συνένεση υπάρχει και για την ρύθμιση και άλλων θεμάτων όπως διαχειρίσεως διαμεθοριακών αξιώσεων. Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Κομισιόν ήταν η οργάνωση δεύτερης ε, διάσκεψης των ενδιαφερομένων μερών, όπου περιγράφηκαν καλύτερα τα θέματα που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτη. Κατέστη σαφές ωστόσο ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά και ιδίω όσον αφορά τον καθορισμό των ποσών της, των αποζημιώσεων. Αυτές οι δράσεις επιτρέπουν στην Κομισιόν να κατανοήσει καλύτερα πού μπορεί να προσφέρει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σε αυτούς, μάλλον τους τομείς θα τους περιλάβει σε μελλοντική ανακοίνωση. Η Κομισιόν ελπίζει ότι η ανακοίνωση αυτή θα ενισχύσει τον διαθεσμικό διάλογο καθώς και την συζήτηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τα θύματα ενδεχομένων ατυχημάτων μέχρι και τους ασφαλιστές. Συζήτηση ουσιώδης για να δημιουργηθεί η απαραίτητη ευρεία συνένεση που θα χρειαστεί να υπάρχει για οποιαδήποτε περαιτέρω πρωτοβουλία που θα βασιστεί στο άρθρο 98 της Συνθήκης Ευρατών. Εν συμπεράσματι θα ήθελα να πω στα αξιότιμα μέλη αλλά και στους αναφερομένους ότι η συζήτηση συνεχίζεται, ότι η Κομισιόν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να λάβει και περαιτέρω μέτρα πέραν της ανακοινώσεως που σχεδιάζει να δημοσιεύσει προσεχώς. Ευχαριστώ. Now, Mr. Becker. Τώρα εσείς κύριε Μπέκερ, αλλά μόνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για ένα λεπτό, ναι. Προβαίνω σε μια διαπίστωση. Την θετική δηλαδή αντίδραση της Κομισιόν ως εξής. Πρόκειται για το αληθινό κόστος των ασφαλίσεων για αποζημιώσεις τρίτων. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της ως έχουσα την ε, αρμοδιότητα να υποβάλει νομοθετικές πρωτοβουλίες, να αρθεί στο των περιστάσεων και να κάνει σωστές προτάσεις. Ευχαριστώ. Τελικώς ε, καταφέραμε να εξετάσουμε κοινώ ε, τις δύο αναφορές. Τις ε, συνοψίσαμε και οι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο αναφέρθηκαν και στις δύο. Συμφωνώ με τον κύριο Μπέκερ για τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά την έκκληση του κυρίου Μπέκερ, νομίζω ότι εν αναμονή μπορούμε να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δούμε τι μέλη γενέστε. Ε, άλλωστε, εμείς ε, όταν δηλώσαμε παραδεκτά τα ε, δύο αιτήματα, ζητήσαμε και γνωμοδότηση της, Ευρωπαϊκής, συγγνώμη, της Επιτροπής Ήτρε. Επομένως, περιμένουμε η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή να μας δώσει κάποια στοιχεία για το στάδιο των δραστηριοτήτων ε, που γίνονται ε, και την άποψή της. Θεωρώ λοιπόν ότι για τις δύο αυτές αναφορές θα πρέπει να μείνουν ανοιχτές ώστε να μπορέσουμε ε, να ε, καταλήξουμε σε αποτέλεσμα μετά τα όσα θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ευχαριστήσω λοιπόν και ε, τους αναφόροντες και όσους με τις υπογραφές τους ε, υποστήριξαν τα θέματα αυτά, διότι έθεσαν ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα αναλάβει η Επιτροπή Αναφορών και θα προσπαθήσει ε, να υπάρχει συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μένουν λοιπόν ανεκτές οι δύο διαδικασίες και περνάμε στην υπαριθμό 24 ε, ενός ε, Γερμανού υπηκόου σχετικά με την επέκταση του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Τέμελιν της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν, επομένως για τη συγκεκριμένη αναφορά δίνω απευθείας το, ρόλο, το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση αυτής της αναφοράς είναι ότι ε, δεν έχει ακόμα περατωθεί η διαδικασία έγκρισης των δύο έργων. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε συμπεράσματα όσον αφορά την εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περίπτωση στην οποία παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και όταν ε, και εφόσον ε, προχωρήσει η διαδικασία ε, υλοποίησης των έργων, θα δούμε κατά πόσον πληρούνται οι προποθέσεις και αναλόγω θα δράσουμε. Έλαβα βέβαια και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αναφέροντα, επομένω θα προσπαθήσω να. Α, μάλλον, συγγνώμη, από τον κύριο Γιάρ και θα προσπαθήσω να τα καλύψω αυτά. Είναι αλήθεια ότι έγινε μια συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των Τσεχικών Αρχών. Αυτό δεν είχε σχέση με τον ε, σταθμό του Τέμελιν, αλλά αφορούσε κυρίω ε, την εφαρμογή τη οδηγία πλαίσιο εν γέννη. Στη συνεδρίαση αυτή όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την ανάγκη η τσεχική δημοκρατία να σεβαστεί τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία στις ε, περιπτώσεις αυτές και κυρίως την οδηγία ε, για ε, πλαίσιο για τα ύδατα. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα και τα διαδικαστικά στοιχεία στα οποία αναφέρεται ο κύριος Γιάρ, αυτά δεν έχουν σταλεί ακόμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επομένως δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη αυτών των ε, τσεχικών εγγράφων και αυτό είναι ε, κάτι το οποίο είναι λογικό σε αυτό το στάδιο γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ολοκληρώνοντας λοιπόν να σας πω ότι παρακολουθούμε ε, προσεκτικά την υπόθεση αυτή, θα δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία διαδότησης και θα σας ενημερώσουμε. vielen Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιθυμώ να σημειώσω εδώ ότι επανερχόμαστε σε ένα βασικό πρόβλημα όπου βεβαίως έχει δίκιο η Κομισιόν ότι όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων δεν θεωρεί ότι υπάρχει αφορμή να εξετάσει αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις διότι η διαδικασία συνεχίζεται. Μπορεί να πει κανείς βέβαια από την άλλη μεριά ότι ευτυχώς εδώ πρόκειται για μέγα έργο και ότι εφόσον ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων μπορεί την επόμενη στιγμή να εξεταστεί και να δουν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αντικτύπου ή να δει αν υπάρχουν άλλες παραβιάσεις. Θα παρακαλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάποια στιγμή το έργο θα έχει δημιουργηθεί θα είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να υπάρξουν απορρίψεις. Γνωρίζουμε ότι βεβαίως υπάρχουν και άλλα σχετικά έργα. Ολοκληρώνεται η διαδικασία διοδοτήσεως και την επόμενη μέρα οι ανεμογεννήτριες ήδη βρίσκονται ε, τοποθετημένες. Και μετά βέβαια ναι μπορούν να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις στους ε, θυγωμένους. Τώρα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνήσει και πει ότι το παρακολουθεί και δεύτερον όταν θα ολοκληρωθεί η φάση του σχεδιασμού θα επανέλθουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι η αρμόζουσα απάντηση για την ώρα και να μην λησμονούμε ότι ένα σημαντικό θέμα είναι και η οδηγία προστασίας των νερών. Ο Μολδάβας γίνεται στον Έλβα, ο Έλβας είναι περιοχή προστατευόμενη Άλλο λοιπόν είναι να ρηπάνει κάποιο επειδή καλλιεργεί ένα χωραφάκι κοντά στον Έλβα και άλλο είναι ένα μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, κρατούμε ανοιχτή την αναφορά και συνεχίζουμε την παρακολούθηση της διαδικασίας. Και θα παρακαλέσω εγώ τον αναφερόμενό μου, εάν ακούσει κάτι που ε, μπορεί να μας ενδιαφέρει, να μας ενημερώσει τάχιστα. Η κυρία Όκεν, κατάλαβα καλά ότι είναι το ίδιο δύσκολο να διαλυθεί μια ανεμογεννήτρια, να αφαιρεθεί μια ανεμογεννήτρια όπως ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Γεια, όχι. Έχουμε όμως το εξή πρόβλημα. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για, τον, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, δείχνουμε εμπιστοσύνη στη χώρα μέλος. Εφόσον ολοκληρωθεί και υποβληθούν παράπονα, ε, δεν κάνουμε τίποτα. Αν όμως υποβληθούν παράπονα, μάλλον όταν ολοκληρωθεί το έργο, τότε μπορούμε να πάμε να εξετάσουμε. Όμως, αυτό που εννοώ εγώ είναι ότι για τις ανεμογεννήτριες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ε, μελέτης αντικτύπου περιβαλλοντικού και τα και δοθούν οι άδειες, την επόμενη μέρα είναι και όλα κατεστημένες. Βέβαια, η ανεμογεννήτρια όμως εύκολο να διαλυθεί. Ακόμα και μια θερινή κατοικία μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί, να γκρεμιστεί. Πολύ λιγότερο όμως από ένα ε, πυρηνικό σταθμό. Ε, ασυνήθιστη αντιπαράθεση στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Γιάρ με την κυρία Όκεν δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο. Δεν ξέρω, ζήτησε κάποιο το λόγο. Κυρία Όκεν, μήπως μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο σας. Όχι, απλώς παρακολουθούσα τις εξελίξεις. Να σας πω το εξής. Όταν συζητήσουμε το δυσάρεστο θέμα ε, ε, της ανεμογεννήτριας, ένα από τα θέματα τα οποία προέκυψε είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο ε, να παροπλήσουμε μια ανεμόνοβη γεννήτρια είναι ίσως το πιο εύκολο πράγμα από πλευράς ενέργειας και ένα από τα πιο δύσκολα είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Είναι σαν να έχετε ένα ποντίκι και, ε, και μια τίγρη. Νομίζω ότι ε, έχουμε ξεφύγει λίγο από το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Ε, το θέμα το οποίο ανακύπτει συνεχώς στην Επιτροπή μας είναι συνήθως ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο είναι στη διαδικασία κατασκευής του και ακόμα είναι ένα αναμονή της αδειοδότησης. Είναι ένα αναμονή λοιπόν της διαδικασίας για να ε, δοθεί άδεια ε, και περιμένουμε την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνήθως λοιπόν ο αναφέρον ο οποίος ε, απευθύνεται σε εμά εκφράζει την ανησυχία τους γιατί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου. Και συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απαντά ότι δεν μπορεί παρά να παρακολουθεί την κατάσταση εν αναμονή της ε, περάτωσης της διαδικασίας. Διότι το πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά αυτή στιγμή όταν ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ε, σωστή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και εδώ νομίζω είναι και το θέμα επί του οποίου συζητήσαμε αρκετές φορές και γι' αυτό ακριβώς και συμμετέχουμε ενεργά στις συζητήσεις για την ε, οδηγία η οποία οδήγησε, και αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και μερικώς δική μας επιτυχία, ε, στο να συμπεριληφθεί στην οδηγία και δυνατότητα προληπτικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κάποια σοβαρά ε, στοιχεία τα οποία ε, προκύπτουν από τη διαδικασία έγκρισης, αδειοδότησης. Η οδηγία βέβαια ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή υπάρχει ο χρόνος μεταφοράς της οδηγίας, επομένως ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις, ε, τους παλιούς τρόπους. Ε, απάντησης. Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να ακολουθήσουμε λοιπόν την πρόταση του συναδέλφου Γιάρ, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα ε, δούμε στο τέλος κατά πόσον οι κίνδυνοι οι οποίοι αναφέρθηκαν από τον αναφερόμενο ε, υπάρχουν και εάν τότε μπορούμε να ζητήσουμε και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διορθωθεί η κατάσταση. Επειδή δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο, νομίζω ότι ακόμα και αυτό θα πρέπει να το ε, αφήσουμε ανοιχτό για να μπορέσουμε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα παρακολουθήσουμε τις δραστηριότητες για να δράσουμε. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει να έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω ούτως ή άλλως τον αναφερόμενο και να περάσω στην επόμενη αναφορά την 2383 το 2013 από τον Heinz Μούτσεκ, αυστριακό υπηκό εξ ονόματος του Μίτερα Βάιντεν Σίδλου Χίρστέτεν, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή επέκτασης αυτοκινητοδρόμου στα προάστρια της Βιέννης και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εδώ έχουμε παρουσία του αναφέροντος. Είναι εδώ λοιπόν ο κύριος Χάιντς Μούντσεκ, στον οποίο δίνω το λόγο για 5 λεπτά για να μας παρουσιάσει την αναφορά του. un momento organizzativo. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, καθώς και εσείς οι υπόλοιποι παρόντες, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λέγομαι Χάιντς Μούτσεκ, δίπλα μου Μπέναρ Σάντλ και ο Αλφες Μπέντερ. Είμαστε εκπρόσωποι πρωτοβουλίας πολιτών στην ε, Κάτω Αυστρία και έχουμε μια αναφορά την οποία επιθυμούμε να σας παρουσιάζουμε και με επιτρέψτε μου να περάσω το μικρόφωνο στον ε, διπλανό μου. Δεν μας ακούν οι δημοτικές αρχές της Βιέννης. Στο έργο που θέλουμε να παρουσιάσουμε πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στο βορειοανατολικό μέρος της ε, Αυστρίας που πιάνει και ύπεθρο αλλά και αστικό χώρο. Δεν είναι βιώσιμο το έργο αυτό και κυρίως θέλουμε να τονίσουμε εδώ παραβιάσεις κατά τη γνώμη μας ευρωπαϊκού δικαίου εκπροσωπούμε 15 πρωτοβουλίες πολιτών στην Βιέννη και περιλαμβάνουν και άλλες εκτός Βιέννης. Εκπροσωπούμε κυρίως τα παιδιά και τα εγγόνια μας που ακόμα δεν ψηφίζουν και που θα υποστούν αργότερα τις συνέπειες από το έργο αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη συμμετοχής των πολιτών εν προκειμένου, που ωστόσο έχει ρυθμιστεί στην ε, σύμβαση του Άρχους, που θεωρούμε ότι δεν τηρείται εν προκειμένου. Δεν έχει υπάρξει διαβούλευση με, τον, με το κοινό σε μια περίοδο όπου έπρεπε να έχει γίνει, όπως προβλέπεται και από την σύμβαση του Άρχους. Όπως είπα και πριν, επιτόπου με τις τοπικές μας αναφορές δεν εισακουστήκαμε, μας απέπεμψαν χωρίς να μας ακούσουν ποτέ. Δεν έλαβαν καν υπόψη τις προηγηθήσεις μελέτες περιβαλλοντικής ανεκτότητας. Για την οδό που είναι μέρος του έργου έχει γίνει συμμετοχή πολιτών, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είχε άλλο παρά διακοσμητικό χαρακτήρα, διότι ούτε η τροχιά της, ε, η διαδρομή δηλαδή της οδού, ούτε τίποτε άλλο δεν συζητήθηκε. Δεν υπήρχαν δηλαδή εναλλακτικές επιλογές, ούτε συζήτηση πραγματική και αντιπαράθεση. Να δώσω τώρα το λόγο, αν με επιτρέπετε, στον άλλο μου ε, παρακαθήμενο, ο οποίος θα εξηγήσει περισσότερα για την στρατηγική. Η συνολική στρατηγική μελέτη των αντικτύπου στο περιβάλλον, στο περιβάλλον έχει παραμεληθεί μέχρι τώρα. Έχει παραληφθεί μέχρι τώρα. Εμείς όμως θεωρούμε ότι αυτή είναι απαραίτητη σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οδηγία Habitat, οικοτόπων δηλαδή, καθώς και το υπόλοιπο κείμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θα το εξηγήσω και με το σχέδιο που βλέπετε. Θεωρούμε επίσης ότι ο δρόμος που έχει ε, σχεδιαστεί επίσης δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Υπάρχει και σε άλλη περίπτωση βέβαια, όχι τούτη εδώ, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι τέτοιε περιπτώσεις είναι παραβιάσει καθαρέ του ευρωπαϊκού δικαίου. Το σχέδιο που βλέπετε στη διαφάνεια δείχνει ολόκληρο το έργο. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Οι πράσινες επιφάνειες που βλέπετε είναι προστατευόμενα, προστατευόμενοι οικότοποι Natura 2000. Εκεί ο μικρός κόκκινος κύκλος είναι βιότοπος ενός είδους νηφίτσας το οποίο είναι προστατευόμενο είδος κατά την αυστριακή νομοθεσία. Βλέπετε ε, μεγάλες αστικές τοποθεσίες, προβλέπετε εκεί ε, οικισμός 20.000 κατοίκων που βρίσκεται υπό σχεδιασμό. Η πράσινη γραμμή είναι ε, σιδηροδρομική οδός διπλής κατευθύνσεως που προέρχεται από την Πρατισλάβα και οι χρωματιστές γραμμές που δείχνω τώρα είναι, ε, υποτίθεται ότι παρουσιάζουν τον σχεδιασμένο δρόμο. Στο σύνολό του, κατά τη γνώμη μας, λόγω του μεγέθους του έργου, είναι απαραίτητο να γίνει στρατηγική ε, μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον, που δεν έχει γίνει όμως μέχρι τώρα. Γκρίζο εδώ είναι, είναι ο αυτοκινητόδρομος που περνάει μέσα από τη Βιέννη αυτοκινητόδρομος που ανήκει στο δίκτυο TEN. Ε, και επίσης ένα τμήμα αστικής οδού που περνά και εισέρχεται μετά σε ένα αυτοκινητόδρομο, εκεί βλέπετε αυτά είναι τμήματα αυτοκινητοδρόμων. Τα νούμερα ε, είναι σημαντικό να εξηγήσω ότι για να μπορέσει να εγκριθεί το έργο το τμήμα αυτό εδώ χωρίστηκε από τον αυτοκινητόδρομο, το 2011 αποφασίστηκε αυτό. Το τμήμα αυτό είναι αυτοκινητόδρομος με τετραπλές λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, χωρίς όμως βοηθητική λωρίδα. Είναι στην ουσία αυτοκινητόδρομος δηλαδή, αλλά μόνο λόγω της έλλειψης λωρίδας εξασφαλίζουν νομοθετικά ότι δεν θα χρειαστεί πλήρης μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον. Εμείς ισχυριζόμεθα και ότι είναι συνολικό σχέδιο αυτό και επομένως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πρέπει να γίνει πλήρη στρατηγικό σχεδιασμός και μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον με συμμετοχή του θυγωμένου πληθυσμού. Εκεί θεωρούμε εμείς ότι έχει γίνει η παραβίαση του δικαίου. Να μου επιτρέψετε να παραδώσω πάλι στον κύριο Μούτσοκ για θέματα ε, του ατμοσφαιρικού αέρα. Όσον αφορά τα σωματίδια ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης έχουμε διαρκώς υπέρβαση των ορίων και στο PMC και στο PMC 2,5 που σημαίνει ότι και στο μέλλον δεν θα μπορούν να επιτυγχάνονται οι τιμές που έχει δεσπίσει ε, το 2015 η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε τακτικές υπερβάσεις των ορίων σωματιδίων ε, σκόνης στον ατμοσφαιρικό αέρα. Μιλούμε για μια κατάσταση σε μια περιοχή όπου ήδη υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και αυτά θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο με τους σχεδιαζόμενους αυτοκινητοδρόμους. Το Ευρωπαϊκό Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει συντάξει μελέτη και έχει περιλάβει το εξής. Τα μέχρι τώρα εφαρμοσμένα μέτρα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη τήρηση των ορίων σε ολόκληρη την Ομοσπονδιακή Επικράτεια του Αυστριακού κράτους. Συνεχίζει στο βορειοανατολικό μέρος της Αυστρίας οι διαμεθοριακές μεταφορές με βαρέα οχήματα από αυτοκινητοδρόμους στην, συμβάλλουν μάλλον στην ε, περαιτέρω ρήπανση. Βλέπετε και αυτό το σχεδόν αυτονόητο ε, γράφημα. Οι κίτρινες στήλε αποτελούν υπερβάσεις των ορίων καθημερινές. Τις βλέπουμε δηλαδή καθημερινά το χειμερινό εξάμεινο. Και αν δείτε και την πράσινη γραμμή πάνω-πάνω, όπου δείχνει το όριο Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015 βλέπετε ότι στην περιοχή μας και στο PM2,5 έχουμε και εκεί σημαντικές υπερβάσεις των ορίων. Συνοψίζω τώρα, εμείς θεωρούμε ότι παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο με την έλλειψη συμμετοχής των πολιτών, με καταστροφή βιοτόπων προστατευομένων ειδών, λόγω έλλειψης της ε, εκτεταμένης στρατηγικής σχεδίασης, ανεπαρκούς αδειοδότησης του έργου και λόγω μη τήρησης των ορίων των ε, σωματιδίων. Υπάρχει και μεγάλη και ιδιαίτερα επίγον χαρακτήρας, διότι έχουν αρχίσει να τρέχουν οι προθεσμίες και γι' αυτό σας παρακαλούμε να ζητούμε μάλλον την υποστήριξή σας και εξέταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Σα ευχαριστώ. Äh, äh, ευχαριστώ, λέει um, Yes, many thanks, uh, Chairman, and thank you also. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τον αναφέροντα. Μόλις τον περασμένο μήνα λάβαμε την αναφορά. Οπότε ακόμα βρισκόμαστε στη φάση της αξιολόγησης. Με μεγάλη προσοχή εξετάζουμε τις πληροφορίες που μας έχει παράσχει ο αναφέραν. Επίσης θα λάβουμε ε, υπόψη και όσα είπατε σήμερα και την όλη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή. Μόλις ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση, τότε θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε την Επιτροπή Αναφορών για το που καταλήξαμε μέσα σε ολίγες εβδομάδες. Η Πρόεδρος. Εσείς κύριε Μπέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εσείς αξιότιμη κύριε αναφερόμενη. Θα είμαι σύντομος. Χωρίς αμφιβολία αντιμετωπίζουμε μομφές σοβαρότατων παραβιάσεων ευρωπαϊκών κανόνων. Χρειάζεται με κάθε σοβαρότητα και ένταση να εξεταστούν οι καταγγελίες αυτές. Το αίτημα απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιληφθούν και μελέτες για ενδεχόμενη προσφυγή. Αναφέρομαι σε ένα θέμα μονάχα. Το ski το Μέλα όπου ένα μόνο θέμα, σε ένα μόνο θέμα μάλλον, κρίθηκε ότι διαχωρισμός του έργου σε τμήματα για να καταστραγηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες οφείλει να οδηγήσει σε απόρριψη συνολικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάρ. Φαίνεται ότι για την Αυστρία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδοτήσεων. Άρα τώρα μπορεί να παρέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακαλώ να δραστηριοποιηθεί ταχύτατα για να μην βρεθούμε πρώτε τελεσμένων γεγονότων. Και οφείλω να συμφωνήσω με τον κύριο Μπέκερ γιατί αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι τελικά είναι αυστριακή σπεσιαλιτέ. Ότι όταν δεν χωράει δηλαδή στα προβλεπόμενα από τον νόμο ένα έργο, το σπάμε σε κομμάτια για να μπορέσουμε να καταστρατηγήσουμε τον νόμο και να μπορέσει, ναι, βέβαια αυτά τα λέω ως μη ειδήμων, από ολόκληρο το έργο αυτό, αφαιρούν α πούμε το εισαγωγικών ένα κομμάτι αυτοκινητόδρομο για να εγκριθεί πιο εύκολα το έργο. Στην ουσία όμως θα διευκολυνθεί η κυκλοφορία και άρα θα αυξηθεί και άρα η ρήπανση θα αυξηθεί επίσης. Έτσι λοιπόν απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην χάσετε χρόνο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους αναφερομένους που ήρθαν και μέχρι τις Βρυξέλλες γιατί έτσι μπορούμε να σας γνωρίσουμε και προσωπικά. Έχετε τώρα τον συνομιλητή σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτως ή άλλως έχετε εμάς ως συνομιλητές που συμπαρατασσόμεθα με τους πολίτες, αλλά έχετε και τον συνομιλητή της Κομισιόν και μπορείτε να έρχεστε, έρχεστε σε επαφή μαζί του εφόσον διαπιστώνετε και άλλα προς καταγγελία. Όμως, έχετε υπόψη σας ότι αν αρχίσει η κατασκευή του έργου είναι πολύ δύσκολο πλέον να αντιστραφεί η ροή του ποταμού. Έχουμε αλλάξει ορισμένα πράγματα το περιβαλλοντικό δίκαιο ακριβώς για να αποφευθούν αυτές οι ελλείψεις γιατί εμείς θέλουμε ήδη από την φάση του σχεδιασμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να παρεμβαίνει ρυθμιστικά όταν διαπιστώνει ελλείψεις. Δεν έχει γίνει ακόμη αυτό, αλλά στην περίπτωσή σας θα πρέπει να γίνει και μάλιστα όσο γίνεται γρηγορότερα. Μια στιγμή λέει η πρόεδρος. Άλλος κανείς από τα μέλη. Οκ, okay, εσείς τότε. Δευτερολογείτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για, την, ε, για, την, για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και επίσης να ευχαριστήσω που υπάρχει η Επιτροπή Αναφορών διότι πρόκειται για θαυμάσιο μέσον της άμεσης δημοκρατίας που είναι τόσο χρήσιμο για να εξηγήσει στον Ευρωπαίο πολίτη ότι στις Βρυξέλλες τον ακούνε. Σας ευχαριστώ για τον έπαινο και την θετική κρίση σας για την Επιτροπή Αναφορών. Η συγκεκριμένη αναφορά μένει σίγουρα ανοιχτή, δεδομένη και της απάντησης της Επιτροπής. ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει και την έκκληση ε, του κυρίου Γιάρ ε, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Εν τω μεταξύ ε, νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν για να συνεργαστούμε σε αυτή τη διαδικασία της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ρωτήσουμε και εμείς απευθείας τις αυστριακές αρχές και μάλιστα τον Υπουργό Περιβάλλοντος για να ζητήσουμε πληροφορίες ε, τις οποίες θα μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε με τις πληροφορίες που μας έδωσαν ε, οι αναφέροντες στη διάρκεια της παρέμβασής τους. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, αφήνουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και ε, θα ζητήσουμε απευθείας και από τις αυστριακές αρχές να μας απαντήσουν για τα όσα ε, μας είπαν ε, τις ανησυχίες δηλαδή των αναφερόντων. Ωραία, σας ευχαριστώ και πάλι για την αναφορά σας. Και περνάμε στο επόμενο σημείο. Αναφορά 0559 του 2009 του Χωσέ Βάθκεθ Γκόμεθ, Ισπανικής Ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή διακλάδωσης αυτοκινητοδρόμου που θα υποβαθμίσει ένα πάρκο στη Σεβίλη. Είναι εδώ ο αναφέρον, ή μάλλον εξ ονόματος του αναφερομένου, ο κύριος Ζήλ Καράσκο, στον οποίο δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Sí. Ε, bueno, mi nombre es Alejandro Gil Carrasco. Alejandro Gil Carrasco ονομάζομαι και εκπροσωπώ αυτό το, το κίνημα για το προστασία του πάρου του, Ταμαργίλια και δίνουμε τη μάχη ώστε να μην κατασκευαστεί αυτό ο δρόμο ύλης ταχύτητας θα περάσει από αυτό το πάρκο πρώτα πρώτα θέλουμε να σας πούμε δύο λόγια τι είναι αυτό το πάρκο βλέπετε εδώ πέρα στην οθόνη είναι αυτή η μέσα στο, στις μπλε γραμμές βρίσκεται σε, κοντά σε αυτή την ε, εργατική συνοικία γύρω από την ε, Σεβίλη και θέλουμε να δώσουμε τη μάχη να προστατεύσουμε αυτόν τον δημόσιο χώρο που ωφελεί την πόλη. γιατί εκτός από πάρκο είναι και αγροβιότοπο. Προστατευμένος ε, καλύπτεται από το, από το μητρό του, το πρωτόκολλο των προστατευμένων πάρκων της ε, Ανταλουσίας ε, για χλωρίδα και πανίδα και εδώ υπάρχουν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορες εποχές και από την Ρωμαϊκή εποχή. Και εδώ είναι παράδειγμα προς μίμηση της συμμετοχής των πολιτών σε ένα έργο, γιατί σχεδόν όλοι οι που και εκεί κοντά ε, συμμετέσχε εις ε, την διαμόρφωση του, του πάρκου και γι' αυτό και όλοι αυτοί που προσχωρήσαν στην κίνηση μας. Τι συμβαίνει τώρα με αυτό το πάρκο. Κινδυνεύει δεν φαίνεται πολύ καλά στην οθόνη, αλλά αν θέλει κανείς να... Αυτό το οποίο θέλουν είναι να περάσουν σε κάποιο, με κάποια κλίση, σε κάποιο άλλο επίπεδο πάνω από το, το, το, το πάρκο, ε, αυτός ο αυτοκινητόδρομος, το πρώτο της που λέγεται, ε, που θα είναι τμήμα του περιφερειακού της ε, Σεβίλης, χωρίς κάποια απογέφερα, και θα αποτελέσει τμήμα της ε, ανάπτυξης αυτής της περιοχής της απειλής που ήταν κάπως ε, παραμελημένη. Βλέπετε κάπου δεξιά, θέλουν να φτιάξουν ένα IKEA, ένα εμπορικό κέντρο και τη εκεί θα, θα και και βιομηχανική ζώνη. Πώς έχει σήμερα η κατάσταση στο πάρκο. Όπως σας είπα, είναι, έχει εκεί πράσινο, είναι, ε, είναι οικότοπος, είναι υγροβιότοπος, Έχουμε πάρα πολλά είδη προστατευόμενα από το Habitat, τη ειδική οδηγία δηλαδή για ψυχότοπους. Επίσης είναι φυσικό περιβάλλον, δημόσιο. Ε, αυτό οφείλει πάρα πολύ και την γειτονιά αυτή που έχει 50% ανέργους. Και επίσης αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το 2006. Τότε σχεδιάσαμε να περάσει αυτός ο δρόμος υψηλής ταχύτητας. Δεν είναι όσο πρέπει να κάνουν από την περιφερειακή κυβέρνηση και από τις δημοτικές αρχές. Παρακάμψαν τις ε, διατάξεις για την προστασία της υπέθρου, θέλουν να φτιάξουν λοιπόν σε αυτό το εμπορικό κέντρο. σχεδιάσαμε αυτήν την διακλάδωση. Παρουσιάζονται πάντως κάποιες εναλλακτικές από το αρχικό σχέδιο. Και εμείς το το θέμα στην Επιτροπή, ήρθε η Επιτροπή σε επαφή με τις τοπικές αρχές, οπότε είπαμε ότι πρόκειται περί παράνομης ε, κατασκευής βάσει της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των πάρκων. Εμείς δρούμε τοπικά επίσης και επικαλούμεθα και ευρωπαϊκές διατάξεις ότι δηλαδή αυτή η διακλάδωση για τον αυτοκινητόδρομο δεν πέρασε ε, από τη φάση της ε, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προβλέπει σχετική κοινοτική οδηγία. Το 2000 έγινε μια σχετική μελέτη αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι άρτια. Τώρα όσον αφορά την επιχειρηματολογία που επικαλούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές λένε, ό, όσα λένε τέλο πάντων είναι έολα επί τη βάση της νομοθεσίας για τη χωροταξία, των πόλεων στην Ανδαλουσία, δεν στέκουν αυτά τα οποία επικαλούνται. Δεν χρειάζεται να γίνει ε, εκεί, ε, να περάσει από εκεί, να γίνει εκεί αυτή η διακλάδωση να περάσει από εκεί ο αυτοκινητόδρομος. Επίσης, αν φτιάξουμε το αυτοκινητόδρομο, θα ματιωθούν όλες τις προσπάθειες που γίνονται το 1996, ούτως ώστε αυτό το πάρκο να μην είναι ε, ε, ένας τόπος ε, χέρσος. και θα υποβαθμιστούν όλες οι ζώνες, οι όμορες του πάρκου. Και έχουμε διάφορε οικολογικέ οργανώσει που συμπλέουν με εμά, οι οργανώσει γυναικείε, Greenpeace, Επίσης έχει κατασκευαστεί αυτό το πάρκο ε, με κοινοτικά χρήματα από το ΦΕΝΤΕΡ, το ΕΡΕΤΠΑ δηλαδή. Είχαν δώσει 22 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πάρκο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά μέσα τώρα θα πάνε στράφη. Θα χωριστεί στα δύο το πάρκο, το κόψει στα δύο αυτοκινητόδρομος πάνε επενδύσεις επομένω οι οποίες ε, έγιναν εκεί. Έχει κατακλείδη να σας αναφέρω ότι το κίνημά μας για το πάρκο Ταμογγίγιο από το 2009 οπότε ξεκίνησαν οι κινήσεις για να φτιαχτεί αυτή η διακλάδωση εμείς αρχίσαμε τις αναφορές έχουμε υποστεί απειλές ε, σωματικής βίας πολιτική δίωξη από τις αρχές της πόλεως της ε, Σεβίλης και από πλευρά τη περιφερειακή ε, διοίκηση. Περιόρισαν το φθόν τι εκδηλώσει μα, ε, μα έκλεισαν ε, τι εγκαταστάσει. Και επίσης ήταν τέτοια αντιπαράθεση με τις αρχές της ε, χωροταξίας της πόλης. Οπότε, αυτό το σχέδιο θεωρούμε για τους λόγους που αναφέραμε ότι είναι παράνομο. Επίσης, ήρθαμε σε επαφή με βουλευτέ και ευρωβουλευτέ, ούτω ώστε να τεθούν οι σχετικές κοινωνικές ερωτήσεις. Οπότε δεν έχουμε άμεση επαφή. Η μόνη μα επαφή είναι μέσω των μέσων ενημέρωση. Δεν υπάρχει ενημέρωση επαρκή. Είναι, είναι κρυπτό και απαραβίστο τα κάνουν όλα. Οπότε εμεί θέλουμε να κηρυχθεί παράνομα αυτό το σχέδιο. Και να σταματήσουμε όλα αυτά τα οποία τώρα απειλούν το Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος της Επιτροπής, ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, και τον αναφέροντα για την παρουσίασή του, ο οποίος ε, λίγο πολύ αναφέρθηκε στο στόχο της αναφοράς αυτής. Η συγκεκριμένη αναφορά επικεντρώνεται στις πιθανές ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να υπάρξουν λόγω ενός συγκεκριμένου τμήματος ε, αυτού του SE35, ε του αυτοκινητοδρόμου, στο πάρκο της Σεβίλης. Δεν αφορά το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου. το πάρκο ε, είχε λάβει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ακριβώς ε, πρέπει να αναφέρουμε ότι ε, υπήρξε χρηματοδότηση για ε, περιβαλλοντική βελτίωση η οποία χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια σε ποσοστό 75%. Επομένως ναι μεν οι ισπανικές αρχές ε, είχαν αναφέρει ότι ένα τμήμα ε, του πάρκου θα είχε ε, δοθεί για τον αυτοκινητόδρομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία πηγαίνει πολύ πέρα από την αναφορά. Η αναφορά όπως σας είπα ε, αφορά μόνο την ε, κατασκευή του τμήματος που θα περνάει από το πάρκο, ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Και δεν περιορίζεται επίσης ε, στο να επαληθεύσει κατά πόσον και με ποιο τρόπο το έργο αυτό προέβλεπε να δοθεί και κάποιο τμήμα του πάρκου για τον αυτοκινητόδρομο ούτε εξετάζουμε απλώς ε, εάν η εκτέλεση αυτού του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου ε, συνάδει ή όχι με την προηγούμενη χρηματοδότηση ενός ε, πάρκου το οποίο χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο ποσοστό από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κάνουν απλώς και μόνο μία νομική ανάλυση. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στο κατά πόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπει η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο του έργου αυτού. Ε, έχει διάφορες ονομασίες, σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται σε κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, ε, σε κάποιες άλλες φορές ε, δακτύλιος ή σύστημα οδικό SE35 ε πρόκειται για το ίδιο έργο. Θα σας δώσω λοιπόν ε, τα στοιχεία βάσει της έρευνας που έγινε. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπορεί να μην διαθέτουμε και θα μπορούσαν ίσως να αλλάζουν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε εμείς. Βάσει των πληροφοριών που διαθέτουμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με, την, με τον ισχυρισμό ότι το έργο αυτό έτυχε ε, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ευρύτερο σχέδιο της αστικής ανάπτυξης της Εβίλης του 2006. Το έργο κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου ή οδού ταχείας κυκλοφορίας ε, όντως ε, έτυχε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά κατά την άποψή μας η ίδια η φύση του έργου, που είναι ένα έργο αστικής ανάπτυξης, χρήσης δάφους, μορφολογίας, ταξινόμησης της χρήσης των εδαφών και ε, εντοπισμός του τι θα μπορούσε να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή έχει μια τέτοια φύση που δεν επιτρέπει να αξιολογήσουμε αναλυτικά όλα τα σχέδια τα οποία υλοποιούνται βάσει αυτού του έργου. Γι' αυτό ακριβώς και τα αναπτυξιακά έργα θα πρέπει να γίνονται ε, με συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, όταν ε, δούμε το γενικότερο σχέδιο αστικής ανάπτυξης, ε, η αξιολόγηση η οποία γίνεται για το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να γίνει σε τόσο επίπεδο λεπτομέρειας ώστε να μπορέσουμε να δούμε και τι συνέπειες θα υπάρχουν και να υπάρξουν και διορθωτικά μέτρα εάν θεωρηθούν απαραίτητα. Και επιπλέον, προφανώς γίνεται με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε όταν ε, γίνεται η αίτηση για την άδεια. Στη συγκεκριμένη απάντηση, περίπτωση βέβαια, ο SE35 ε ε, φαίνεται ότι προφανώς έχει ε, καταμεριστεί σε διάφορα έργα μέσω των οποίων υποτίθεται ότι θα γίνει το συνολικό μεγαλύτερο έργο. Ακριβώς αυτός ο καταμερισμός και το γεγονός ότι γίνονται μικρότερα κατασκευαστικά έργα σημαίνει ότι η αξιολόγηση γίνεται αργότερα σε κατοπινό στάδιο και όχι στο πρώτη, στην πρώτη φάση. Επομένως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αξιολόγηση που κάνει το έργο μπορεί ε, να διαπιστώσει τι συνέπειες μπορεί να έχει το έργο στο περιβάλλον και σε όλους τους υπόλοιπους ε, ε, παράγοντες που αναφέρει η οδηγία. Πέραν αυτού, εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και με το επιχείρημα βάσει του οποίου το έργο αυτό, αυτό το γενικότερο σύστημα αυτοκινητοδρόμων αν θέλετε, ε, θεωρείται απλώς ένας δρόμος. Και επομένως γίνεται εξέταση απλώς και μόνον ε, κατά πόσο θα πρέπει να εξαιρεθεί ω αυτοκινητόδρομο ή βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπουν το παράρτημα 1 και παράρτημα 2 τη οδηγία, ω έργα τα οποία ε, βάσει της οδηγία θα πρέπει να την χάνουν αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θεωρούμε ότι η ερμηνεία αυτή σε αρκετέ περιπτώσει απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προκύπτει σαφώς ότι η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στα έργα μεταρρύθμισης και στα έργα βελτίωσης ε, του αστικού περιβάλλοντος ε, είτε είναι του παραρτήματος 1 είτε είναι του παραρτήματος 2 όταν έχουν σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον, ε, λόγω του μεγέθους του της, της φύσης τους ή οποιοδήποτε άλλου λόγου, πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. δεν είχαμε σε άλλες περιπτώσεις ε, έργα αντίστοιχη κλίμακας ε, δακτυλίων περιφερειακών ε, επί των οποίων να θεωρήθηκε βάσιμο αυτό το επιχείρημα. Αυτό το επιχείρημα το υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αποφάσεις του δικαστηρίου ήταν τελεσίδικες για το θέμα αυτό. Επομένως, ανακοινώσαμε στις Ισπανικές Αρχές ότι θα ξεκινήσει απευθείας μια διαδικασία επιπαραβάση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τον αναφερόμενο, διότι μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτή την υπόθεση, η οποία είναι πολύ γνωστή. Το συγκεκριμένο πάρκο ε, σημαίνει πολλά ε, το πάρκο Ταμαργίγιο για την Σεβίλη και για ιστορικούς λόγους, αλλά και για να υπάρχει ένας πνεύμονας ε, οξυγόνου μέσα στην πόλη της Εβίλης. Και επίσης οι πολίτες προσπαθούσαν να έχουν ένα φυσικό χώρο, ο οποίος εγκαταλείπεται σιγά σιγά και καταφέραμε πάρα πολλά ε, σε αυτά τα 96 εκτάρια τα οποία περιλαμβάνεται το πάρκο. Υπήρχαν υποδειγματικά προγράμματα ε, δημιουργία σχολικής περιβαλλοντικής συνείδησης για παράδειγμα, κάτι το αποτέλεσε υπόδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο ε, μπόρεσαν να συμμετέχουν οι πολίτες, πάνω από 60.000 οικογένειες, 200.000 μαθητές και εγώ πραγματικά θα χαίρομαι ιδιαίτερα που το θέμα αυτό έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσουμε μια λύση και για να μην επιτρέψουμε να γίνει κάτι το οποίο σίγουρα θα αποτελούσε πολύ σημαντική ε, παρέμβαση σε αυτό το πνεύμα οξυγόνου. Μετά από τα πόσα άκουσα βέβαια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η πρόταση νομίζω είναι να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, αλλά θα ήθελα να αναφέρω και το εξή. Εγώ συμφωνώ απολύτω με τα όσα είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί ε, να παρακάμψει κάποιος την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ανάγκη ε, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς συζητήσαμε με τη Μαδρίτη ε, για το πώς προσπαθούσαν να κοροϊδέψουν για την κατασκευή του Μη 30, ενός δρόμου ο οποίος θα περνάει μέσα από την πόλη και οι τοπικές αρχές τον αποκάλεσαν δρόμο για να μην χρειαστεί να κάνουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε είχε ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση και νομίζω ότι όντως ε, ε, το μόνο που λείπει είναι να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πρόκειται για κοροϊδία οι τοπικές αρχές προσπαθούν να παρακάμψουν ε, μία απέτηση της οδηγίας, ε, να υπάρχουν δηλαδή σε αυτά τα έργα, σε κατασκευές αυτοκινητοδρόμων, υποχρεωτικά ε, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα και χαίρομαι, δεν μας χαροποιεί συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πούμε σαφέστατα ότι είναι υποχρεωτική αυτή η διαδικασία επιπαραβάση και ε, αυτό το οποίο ξεκινά αυτή τη στιγμή κατά της Ισπανίας και πιο συγκεκριμένα κατά του Δήμου της Σεβίλης μας επιτρέπει κάτι σε μελιώδες, δηλαδή τη διατήρηση του πάρκου ε, και να τον προστατέψουμε ενάντια σε αυτές τις επιθετικές πολιτικές που θέλουν να το καταστρέψουν. Ζητώ φυσικά να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τη διαδικασία επιπαραβάση και να λάβουμε και την απάντηση των τοπικών αρχών και φυσικά ο ίδιος ο αναφόρον να μπορεί να δει ε, και η διεισόμαση τι γίνεται με την όλη διοικητική διαδικασία και να έχει και περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιράτσο ευχαριστώ. Συμφωνώ με όλο όσα είπε ο Πιλιμάγερ. Θέλω να σταθώ στην θετική ανταπόκριση από πλευρά Επιτροπή. έχουμε πάρα πολλέ παρόμοιε περιπτώσει μη τήρηση των οδηγιών. Ακούμε σωρία προφάσεων και δικαιολογιών σε αυτή την περίπτωση. όμω ενήργησε με επιμέλεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάλυψε τους αναφέροντες. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά ενημερώθηκα από τον συνάδελφο Μέγερ τι έγινε σε αυτές τις συνοικίες της ε, Σεβίλης. Και θέλω στον αναφέροντα να το πω ότι τον ευχαριστώ για το έργο του. Γιάννης. Θα είμαι σύντομος κυρία Πρόεδρε, γιατί συμφωνώ με τη γνώμη όσων ε, τοποθετήθηκαν προηγουμένως αλλά και με τον αναφέροντα για το πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε και να συμβάλλουμε σε αυτό του είδους το πάρκο το οποίο βοηθάει και το περιβάλλον και αποτελεί και χώρα αναψυχής και ξέρετε ότι είμαι σε Βιλιάνο και όπως είπε και ο κύριος Βιλιμάγερ το ξέρουμε πολύ καλά και το εκτιμούμε αυτό το πάρκο. Πολύ σημαντικό γιατί το ρεμπλάμε και αυτή την περιοχή. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Έχουν δίκιο οι όσο καταγγέλουν. Απλώς δεν, είμαι, δεν δουλεύω εδώ στην Επιτροπή σας ε, και θα πρέπει ίσως να έχουμε καλέσει, δεν μπορεί να σου πω, δεν είμαι τακτικότητα ε, ε, μέρος, αλλά να έχουμε καλέσει εμπλεκόμενες αρχές. Δεν, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά θα έπρεπε να ακουστεί η φωνή της περιφερειακής κυβέρνησης Ανδαλουσίας, αλλά και των δημοτικών αρχών. Ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επίτροπη και όλα αυτά βασίστηκαν σε ανάπτυξη επιχειρημάτων με την έγγραφη διαδικασία. Πέραν αυτό πάντως, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε. Θα πρέπει να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσει το θέμα, όπως τα είπε και ο εκπρόσωπος αυτής. Α, ε, Μα αυτά τα πράγματα τα έχουμε ξαναδεί. Έχουμε ένα αίσθημα του ντεζοβίου ήδη από τις αρχές που ήμουν μέλος της Επιτροπής Αναφορών και είχαμε πάει με αντιπροσωπεία στην Μαδρίτη για να δούμε και πολλοί πολίτες ήταν εκεί παρόντες και η εντύπωση που είχαμε και από τους πολίτες αλλά και από το Δημοτικό Συμβουλίο Μαδρίτης. Ήταν σαφές ότι πρόκειται για αυτοκινητόδρομο. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Αλλά το αποκαλούσαν κάγε, δρόμο δηλαδή. Σαν ήταν δηλαδή δυνατό να αλλάξουν τη φύση ενός μεγάλου πλατιού αυτοκινητόδρομου να γίνει μικρός δρόμος και με τον τρόπο αυτό να αποφύγουν την επιβολή ή την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Βέβαια δεν δεχτήκαμε τα πράγματα αυτά και χρειάστηκε βεβαίως να συγκρατηθούμε, να συγκρατήσουμε τις αυθόρμητες αντιδράσεις μας διότι ήταν τελείως αστείο. Βέβαια και όλοι οι πολίτες είχαν συνεργαστεί και εργαστεί για να γίνει πραγματική μελέτη επιπτώσεων για να γίνουν σεβαστές οι απαιτήσει του νόμου σε μια μεγάλη πόλη όπως η Μαδρίτη. Ευχαριστώ λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν φάνηκαν τόσο κακοί εκείνη τη φορά, αλλά τουλάχιστον τώρα δείχνουν μια ξεκαθαρή και ελπίζω εσείς να φανείτε πιο τυχεροί και πιο επιτυχημένοι. Γιατί αν να περιμένουμε μέχρι ότου γίνουν οι καταστροφές και ο Πέτερ Γιάρ για παράδειγμα, το πώς τον Πέτερ και ο αυτοκινητόδρομος πώς να ξυλωθεί όταν θα έχει φτιαχτεί. Χαίρομαι όμως που λέει η Επιτροπή αυτά που λέει και σας εύχομαι, ε, μάλλον σας ε, βεβαιώνω ότι θα έχετε την υποστήριξη για την υπόθεσή σας που προσπαθείτε να κρατήσετε κάποιο πράσινο στην ε, πόλη της Σεβίλης. Όχι, εγώ δεν είμαι και από την περιοχή, δεν, δεν γνωρίζω από κοντά αυτό το, το, το, πάρκο όπως ο κύριος Μέγερ, ούτε θα τολμούσε όπως ο κύριος Γιάννη, ο οποίο είναι από εκεί που μας επενδύμησε. Όμως, θέλω στον κύριο Μέγερ, που μας μίλησε για τις δημοτικές αρχές της Σεβίλης, ότι ε, έχουμε την αρμόδια αρχή ε, που ασχολήθηκε, που ασχολήθηκε με το περιβάλλον για τον αυτοκινητόδρομο 35 ε, της Σεβίλης αν θυμάμαι καλά, επομένω, η ενωτική αριστερά, το κόμμα του κυρίου Μέγερ, ε, κυριαρχεί μαζί με τους σοσιαλιστές στις ε, περιφερειακές αρχές της ε, Ανταλουσίας. Πάντως, βλέπουμε εδώ στο φάκελο ότι θα διαβάζω για να έχετε υπόψη τι έγινε και πώς έχουν εξελθεί τα πράγματα και λέει ότι σήμερα έχουμε αυτή την υποβολή ε, αυτού, αυτού του, αυτής της διακλάδωσης, οπότε λέει εδώ πέρα ότι σε αυτή τη, γίνεται αυτή η, ενημέρωση του κόσμου και έχουμε επομένω ε, αυτόν τον αυτοκινητόδρομο που είναι προς το δημόσιο συμφέρον και ε, το Υπουργείο Υποδομών έχει ενημερώσει τον, ε, τον, τον κόσμο και έχει ε, ημερομηνία Φεβρουάριο του 2014 πρώην μηνός, οπότε και λέμε ότι έχει 29 επιχειρήματα από διάφορες αρχές, διάφορους φορείς που έχουν υποβληθεί σε αυτή την αρχή για τους ε, αυτοκινητοδρόμους και είπε ότι επιβεβαιώνονται οι, οι ευμενείς γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων, συνομοδίων αρχών που έχουν υποβληθεί στο, στις αρχές χωροταξίας ούτως ώστε να εγκριθεί το έργο. Και αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ είναι ότι σε καμία περίπτωση μέχρι εκείνη την ημερομηνία από ό,τι αναφέρεται αυτή η Γενική Διεύθυνση δεν ε, ξεκίνησε την ανάθεση του έργου για κάποιο τμήμα αυτού του δρόμο. Δεν αναφέρεται λοιπόν με τίποτα. Νομίζω εγώ ότι σε κάποια περίοδο υποβολή των, των επιχειρημάτων είναι πάρα πολύ πρόημο. Πρόημο να πούμε ότι ε, έχει το θέμα προχωρήσει ουσιαστικά και άρα θα πρέπει να, να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να δούμε τι κατεύθυνση θα πάρουν τα πράγματα σε σχέση με αυτές τις ε, προτάσεις που όπως προείπα έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία χωροταξίας των Δημοτικών Αρχών της πόλης. Πρόεδρος. Κύριε Μαϊρά. Ήθελα να πω στον κύριο ότι αυτή η επιστολή που μας ε, διάβασε ξεκαθαρίζει το ότι αρμοδιότητα έχουν οι αρχές. Συγκεκριμένα οι αρχές για τις υποδομές, για τα έργα το Υπουργείο Υποδομής συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά, και εγώ και ο κ. Γιάννη θα έχουμε στρατευτεί και έχουμε δεσμευτεί ότι σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για συναρμοδιότητα. Κάποιοι από τι λίγε αρμοδιότητε που έχουν οι περιφερειακέ διοικητικέ αρχέ τη και άρα θα πρέπει ε, και μαζί με, τις, με τα ευρωπαϊκά όργανα στο πλάι αυτών των πολιτών που δίνουν τη μάχη τους. Πολύ σημαντικό για την υπόθεση μου, το ποιος ήταν Διάφορες οργανώσεις, επομένως, επικοινώνησαν με τις αρχές που αναφέρονται στην επιστολή και είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ σε σχέση με την κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου. Και είπαμε ότι υπάρχει παραπληροφόρηση από τις δημοτικές αρχές πέραν το ότι φύγονται τόσες συνοικίες και αυτή η παραπληροφόρηση έχει επιδράσει και στην γνώμη που διαμόρφωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι σήμερα δεν έγινε η επικοινωνία, η ενημέρωση όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. υπάρχει κάποιος υπεύθυνος στο Δημαρχείο της ε, Σεβίλης που ανήκει στο Λαϊκό ακόμα και δεν έχει λάβει υπόψη τις εναλλακτικέ όπως τις έχουμε υποβάλει. Και έχει θεωρηθεί ότι η μόνη λύση είναι το να περάσει πάνω, μέσα από το πάρκο, αυτός ο δρόμος. Γιάννη. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια, αλλά θέλω να συμπληρώσω κάτι κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον στο μέλλον θα καλέσουμε εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφερειακής Διοίκησης. Και όσο είπε ο κύριος Μέγερ. Και όπως είπε και ο κύριος ε, Ιτουργκάιθ, να έχουμε εκπροσώπους του Υπουργείου Έργων Υποδομής που είναι αυτοί που θα έχουν τελευταία λέξη από πλευράς κυβέρνηση της χώρας. Κύριε Τούντα με αυτή την νομοθεσία όπως βλέπουμε δεν έχουμε εδώ αρκετούς βουλευτές. Συζητούμε σε μια μισοάδια αίθουσα. Ε, ίσως γιατί ήρθε τώρα η αναφορά προς συζήτηση λίγο πριν το τέλος της θητείας. Γιατί το λέω αυτό. Ε, ίσως η γραμματεία μας και εσείς επίσης θα πρέπει να, θα πρέπει να φροντίσετε το θέμα να μην κλείσει, να το επαναφέρετε και τότε ε, θα, είμαστε, θα είναι άλλοι βουλευτές εδώ. Είτε γιατί έχει ανανεωθεί ε, η Επιτροπή από Μελών, είτε επειδή εμείς μπορεί να μην είμαστε καν ε, βουλευτές. Σας ευχαριστώ όλους και κυρίως ευχαριστούμε τον αναφερόμενο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα κάνει. Η αναφορά φυσικά θα παραμείνει ανοιχτή, δεδομένου και ότι και εμείς θέλουμε να παρακολουθήσουμε την αλπορία του θέματος για να κάνουμε φυσικά αυτό που μας αναλογεί στη συνέχεια, να φέρουμε δηλαδή τους πολίτες απευθείας σε επαφή με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε μέσω να γράψουμε επιστολή και στις ε, τοπικές αρχές, ώστε να υπάρξει ίσως στο μέλλον και κάποια ακρόαση, να υπάρξει δηλαδή και μία αντιπαράθεση μεταξύ τοπικών αρχών και εκπροσώπων της αναφοράς. Όπως υπενθύμησε βέβαια και ο κύριος Γιάννες, εμείς ε, θα ανοίξουμε την πόρτα για αυτή τη δημοκρατική αντιπαράθεση μεν, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ε, όλα αυτά θα γίνουν από όλους όσους θα είναι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ολοκληρώνεται η συζήτηση τώρα, μένει ανοιχτή η αναφορά και καλούνται οι τοπικές αρχές της Σεβίλης να συμμετέχουν σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε τον αναφέροντα και ευχαριστούμε και τους συναδέλφους. Συνεχίζουμε λοιπόν με το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, αναφορά 0971 κάθετο 2013 του Κάρλο Αλόνσο Θίδα, Ισπανικής Θεσσαγένεια, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στη δεξαμενή Ογιόλα στη χώρα των Βάσκων. Ο λόγος των Χωσέ Χαβιέρ Βάσκες Δολάσκο. Καλησπέρα σα. Κυρίε και κύριοι, καταρχά. η οργάνωσή μας ε, των ε, όσων βρίσκονται γύρω ε, από την δεξαμενή Ογιόλα ε, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε εδώ για να σας αναφέρουμε την κατάσταση του πόσιμου νερού στη δεξαμενή Ογιόλα, το οποίο μολύνεται από μια επικίνδυνη ουσία και ζητάμε τη βοήθειά σας ώστε οι τοπικές αρχές, οι αρχές των αυτόνομων περιοχών και οι ε, κεντρική κυβέρνηση να ε, κάνουν κάτι για το θέμα αυτό. Ζητούμε τη βοήθειά σας και κάνουμε μία έκκληση για να ζητήσουμε να ε, υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, να υπάρξει συμμετοχή και να ακουστούν οι απόψεις όλων όσων πλήττονται από αυτή τη διαδικασία και να αναζητήσουμε λύσεις με τις τοπικές αρχές που εμπλέκονται στο όλο θέμα. Καταρχάς ε, την εταιρεία υδάτων της χώρας των Βάσκων, ε, τους δήμους των ε, περιοχών που πλήττονται και τις αρχές δημόσιας υγείας της χώρας των Βάσκων. Τον Οκτώβριο του 2010 η Mercedes Εστέβες είπε ότι η ουσία αυτή είναι καρκινογόνος και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Ακόμα και αν είναι πολύ μικρά τα ποσοστά, δεν είναι μηδενικά. Υπάρχουν και, άλλους, ε, και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι στην ε, κοινότητά μας να διαχειριστούμε τα θέματα και θα πρέπει να αποφύγουμε περί κινδύνους. Κυρίες και κύριοι, για να σας πω για ποιο λόγο κάνουμε αυτή την αναφορά. Η δεξαμονή της Ογιόλα μετά από αρκετά περιστατικά που είχαμε το 2007 έχει συνδεθεί ε, από τις 22 Απριλίου με περισσότερες περιοχές ε, και εκθέτει αρκετούς ε, ανθρώπους οι οποίοι ζουν στους διαφόρους δήμους ε, του, της περιοχής. Και η εταιρεία υδάτων της χώρας των Βάσκων λέει ότι θα γίνει στη συνέχεια επεξεργασία του νερού, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας όταν εμένει ο κίνδυνος. Μπορεί να γίνει επεξεργασία μόνο με ενεργό άνθρακα. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα καθορίζει σαφώς στόχους και λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη ε, για θέματα ρήπανσης ε, με γνώμονα τη δημόσια υγεία και τη διατήρηση των υποσυστημάτων. Θέλουμε λοιπόν να ληφθεί αυτό υπόψη και το ζητούμε διότι αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη δεξαμηνή υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και στον όλογο ε, της ουσίας αυτής η οποία είναι καρκινογόνος και δεν μετρούνται ε, τα, η, ποσότητα που υπάρχει αναγραμμάρια, υπάρχουν και οι της ουσίας αυτής και πιο συγκεκριμένα υπάρχει το ισομερές δέλτα για το οποίο κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί εάν τα 27 νανογραμμάρια αναλύτρο που λέγεται ότι εφαρμόζονται, εφαρμόζονται όντως. Δεν αναλύεται επίσης η παρουσία της ουσίας αυτής ε, στα ε, λιμνάζοντα ύδατα. Σε όλες αυτά τα χρόνια έγινε μόνο μία μελέτη στη Δεξαμενή το 2009 και κάποια στιγμή καταλήξαμε στο 1.800.000 νανογραμμάρια όπως ε, μπορείτε άλλωστε να αποδείξετε και στην έκθεση την οποία σας έχουμε επισυνάψει στα έγγραφα τα οποία σας δώσαμε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα δράσης για την ε, ε, εξάλληψη της ουσίας αυτής όπως προβλέπει η οδηγία. Δεν υπάρχει μητρό προστατευόμενων περιοχών υδάτων για την παραγωγή πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και επίσης δεν υπάρχουν μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου. Όλα αυτά φυσικά δεν μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε με κατάλληλο τρόπο του κίνδυνου οι οποίοι ανακύπτουν και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο πρόβλημα αυτό ε, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, για τον υδρογονάνθρακα αυτό και θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τα γεγονότα, κυρίως το γεγονός ότι δεν τηρείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την πρόσβαση σε πληροφορίες και δημόσια συμμετοχή σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα ώστε να υποχρεωθεί η Ισπανική κυβέρνηση ε, να διορθώσει αυτές τις ελλείψεις ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως προκύπτουν από την ανάληψη. Ζητούμε επίσης από την Ισπανική κυβέρνηση να εγκρίνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές ε, της αυτόνομης περιοχής της χώρας των Βάσκων και οι δημοτικές αρχές να φροντίσουν να τηρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σε σχέση με τα όσα σας αναφέραμε και θέλουμε να ανασταλεί η χρήση της δεξαμενής ε, ογιόλα για την παραγωγή ποιόσιμου νερού ε, μέχρι να επιβεβαιωθεί η ε, ποιότητα για την υγεία και το περιβάλλον. Και ζητάμε από την Ισπανική κυβέρνηση να εγγυηθούν και το δικαίωμα της πρόσβασης σε πληροφορίες και δημόσια συμμετοχή από πλευράς των ενδιαφερομένων αρχών να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας, διότι δράσεις σαν αυτές είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν εμπιστοσύνη και προσδεθούν και κάποιο νόημα στα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φερνάντο Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε γνώση των όσων ανέφερε ο αναφέρον μέσω μιας αναφοράς η οποία αναφέρθηκε το 2013 ε, και από διάφορες γραπτές ερωτήσεις προς το Ευρωπαϊκό, ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από αυτό ήρθαμε σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση των ουσιών αυτών που περιλαμβάνονται στα ύδατα της δεξαμενής της Ογιόλα και στο πόσιμο νερό το οποίο χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Και επίσης ρωτήσαμε και τι μέτρα λαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση από τις Ισπανικές Αρχές προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα μόλυνσης των υδάτων τα οποία προέκυψαν. Οι πληροφορίες που λάβαμε προς το παρόν αναφέρονται απλώς σε μια μερική ανάλυση της κατάστασης που υπάρχει στη συγκεκριμένη δεξαμενή. Γι' αυτό ακριβώς θεωρήσαμε ότι ε, θα πρέπει να στείλουμε αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες στα πλαίσια του προγράμματος Pilot και αφού ληφθούν όλες αυτές οι πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει ίσως να αποφασίσει ε, για το θέμα αυτό με στόχο να τηρηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω ότι γνωρίζω αρκετά καλά την κατάσταση. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία είναι καταδικασμένοι από τα εργοστάσια τα οποία βρίσκονται στην ε, περιοχή, εργοστάσια τα οποία έκλεισαν στη δεκαετία του 80 και δημιούργησαν προβλήματα όχι μόνο στην περιοχή αλλά σε όλο το βυσκαϊκό κόλπο και πλήττουν ε, μεγάλο τμήμα του βυσκαϊκού κόλπου και το ίδιο οδήγησε και στην έγκριση μιας περιοχής ασφάλειας για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την περιοχή και να μπορέσουμε να καθαρίσουμε από τη μόλυνση. Όσον αφορά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αυτή είναι προφανής διότι υπάρχει κίνδυνος όταν υπάρχουν τόσο πολύ επικίνδυνες και καρκινογόνες ουσίες οι οποίες μεταδίδονται μέσω του πόσιμου νερού και θεωρώ ότι για το θέμα αυτό και η εταιρεία υδάτων ε, του Μπιλμπάο και ε, οι αρμόδιες αρχές θεωρώ ότι μάλλον ασυνείδητα δρούσει, Δεν κάνουν τις ε, κατάλληλες αναλύσεις και δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφύγουν όλοι όσοι καταναλώνουν πόσιμο νερό από τη δεξαμενή αυτή ε, να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θα πρέπει να φροντίσουν το νερό να την χάνει ανάλογη ποιότητα και κατάλληλα μέτρα δεν έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή. Το πόσιμο νερό της δεξαμενής του Ισογιόλα ε, είναι σαφώς κακής ποιότητας, ενώ οι αρχές της κυβέρνησης ε, της χώρας των Βάσκων φαίνεται να αδρανούν για το θέμα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών της περιοχής. Είναι επωνίδιστη αυτή η κατάσταση και θα ήθελα εδώ να ε, καταδικάσω τα όσα συμβαίνουν. Από ό,τι βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει επικαιροποιημένες πληροφορίες για να μπορέσει να αποφανθεί. Ελπίζω ότι οι αρμόδιες αρχές και της χώρας των Βάσκων και οι ε, αρμόδιες τοπικές αρχές, η εταιρεία υδάτων του Μπιλμπάου να μπορέσει να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις και να προσπαθήσουν να αποφύγουν αυτό το κίνδυνο για την δημόσια υγεία, δηλαδή τη χρήση ε, του νερού που έχει μολυνθεί από τη συγκεκριμένη ουσία και ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά εν αναμονή των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας πιθανής λύσης για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ετούντες. Η πρόληψη είναι κάτι το οποίο μα χαρακτηρίζει εδώ ε, όμως από την άλλη μεριά ενεργεί αργά η Ευρώπη και χρειάζονται εδώ πέρα κάποιε εγγύσει όπω λένε οι τούντε, τόσο ώστε όταν κανεί ανοίγει τη βρύση να έχει την εγγύηση τη ασφαλείας ότι δεν θα πίνει νερό βλαπτικό, βλαβερό για την υγεία. Όπω είπε και ο συνάδελφο, το θέμα επήγει, άρα θα πρέπει η επιστολή να διαβάσει. Η επιστολή σε αρμόδιε ε, ε, αρχέ και στην βασική κυβέρνηση και στις διοικητικές αρχές στις ε, οποίες αναφέρθηκε. Δημοτικές αρχές, όλο, όλους τους εμπλεκομένους να διατυπώνουμε εκεί την ανησυχία μας ότι θα πρέπει να κατησχύσει η αρχή της σύνεσης. Άρα, να μας απαντήσουν έτσι τόσο ώστε να έχουμε τις εγγύσεις ότι δηλαδή αυτός ο εγωριότοπος, αυτό το έλος τέλος πάντων δεν θα, ε, καταλήξει σε πόσιμο νερό. Οπότε θα πρέπει αυτό το θέμα να και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν έχω λάβει ακόμα γραπτή απάντηση περί του. όμως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Όλοι θέλουμε ταχεία διεκπαιρέωση. Είναι θέμα δημόσια υγεία, ανθρώπινη υγεία. Δεν μπορεί να περιμένει το θέμα. Α επιταχύνουμε τι ε, ενέργειε του αρμοδίε αρχέ να δώσουμε τι εγγύσει που θέλουν. Κύριε Γκαρθία. Πρώτα πρώτα. Θα πρέπει να τονίσουμε το πόσο αξιόλογη πρωτοβουλία ανέλαβαν οι, ε, αναφέροντες και ο Κάρλος Σιδά Δεν έχω μπορέσει επιτόπου να δω τα, τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία αναφέρθηκαν οι αναφέροντες, αλλά Είχε πάει συνάδελφο η οποία είναι έγκυο τώρα σε προχωρημένη φάση δεν μπορεί να έρθει εδώ. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα ακουστεί η φωνή μας. Διαπιστώσαμε ότι και σε άλλε περιπτώσεις όπως και εν προκειμένου είναι δύσκολο να μας ακούσουν. Να μας ακούσουν και στην Ευρώπη αλλά και επί τόπου εκεί που σοβεί το πρόβλημα. Μέσα στην αρχή τη διαδρομή. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε, να αναλύσουμε τις πληροφορίε όλες αυτές τις οποίες ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για κάποιες περιοχές που γνωρίζω από τη Μαδρίτη μακροπρόθεσμα. Επηρεάζεται η υγεία των κατοίκων εκεί, εκείνοι που μένουν εκεί, αναπνύουν τον αέρα, πίνουν το νερό αυτών των μολυσμένων περιοχών. Άρα, υπάρχει κάθε λόγος να μην έχει αναφορά. Και να δούμε ποιοι είναι πραγματικά οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και τι μέτρα θα ληφθούν. Μιλάμε εδώ για ανθρώπινη υγεία. Άρα πρέπει να δούμε αν είναι εδώ πέρα όντως τρίχη περίπτωση κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Επομένως δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν και να ξανά ευχαριστήσω τον φορέα που έφερε την υπόθεση αυτή στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, το, σώστε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα να προωθήσει την υπόθεση αυτή για να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε τώρα για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Πρέπει να σα πω ότι και από πλευρά του Λαϊκού κόμματο πρόκειται να ζητήσουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και κάτι το οποίο δεν το είπαν στις 23 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο του Μπαρακάλτο εγκρίθηκε ένα ψήφισμα το οποίο το Λαϊκό Κόμμα κατέβασε. Ζητήσαμε να αξιολογηθεί η ποιότητα του πόσιμου νερού της δεξαμενής Ογιόλα. Και συνέπλευσαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του βασικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Να ζητήσουμε την γραμματεία μας, για να συμφωνείτε, να μην ανοιχτεί η αναφορά. Να στείλουμε στην εταιρεία Ιδάτων του Μπιλμπάου την επιστολή, στην διοίκηση της χώρα των Βάσκων, στο, Δήμο του Μπαρακάλδο, στην Ισπανική κυβέρνηση. Και έτσι θα έχουμε τη επαφή με όλους τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Οπότε ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο μέσα διάταξης. Οπότε απομείνει να υπενθυμίσω σε όσους είναι μέλη, όσους είναι συντονιστές μας τέλος πάντων, ότι στις 5.30 θα ε, συνεχίσουμε τη συνεδρίαση οι συντονιστές.